Welcome to everybody. Uh, thank you for being here. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλωσορίζουμε λοιπόν τους φιλοξενούμενους για το Erasmus Plus Καλωσορίζουμε επίσης και τους υπεύθυνους για τη μελέτη η οποία ζητήθηκε από το Policy Department 2, τους κυρίους Κετούναν και Γουότα. Και τώρα θα συνεχίσω στα Ιταλικά. Μπορείτε να ακούσετε τα ακουστικά σας. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας λοιπόν. Σήμερα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα εφαρμογής των προτάσεων γύρω από το Erasmus Plus, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τους νέους, για τη νεότητα για τα πανεπιστήμια και τα λοιπά. 14-20. Έχει ληφθεί μία απόφαση από τη διάσκεψη των Προέδρων η οποία λέγει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί του χρόνου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος το 2017. Κατά κάποιο τρόπο εμείς προκαταλαμβάνουμε αν θέλετε την διαδικασία αυτή για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί μετά τις θεσμικές αλλαγές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περισσότερες ελεγκτικές δραστηριότητες και δεύτερον γιατί θα ήταν ε, πολύ χρήσιμος τελικά ένας τέτοιος τύπος επαλήθευσης έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωρίζει τις προτάσεις μας γύρω από τη διαχείριση του προγράμματος, γύρω από τους στόχους που έχουμε θέσει και να δούμε ακριβώς τι τροποποιήσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν από το 2020. Θα παρουσιαστούν δύο μελέτες. Το πρώτο είναι αξιολόγηση των πρώτων εμπειριών από το Erasmus Plus, από το Academic Operation Association συλλέγει μέσω ερωτηματολογίων στοιχεία και συνεντεύξεων και η δεύτερη μελέτη από την υπηρεσία τεκμηρίωσης είναι το Key Action 2. Χρηστές πρακτικές, ε, ενημέρωση για θέματα που αφορούν την νεότητα έχει συγγραφεί η δεύτερη πρόταση από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου του Τούρκου. Έχουμε εδώ επίσης τον Διευθυντή ε, Βίκε από την Γενική Γραμματεία Νέων στην Γερμανία, τον κύριο Στράτσαρτ από την Αρμόδια Υπηρεσία της Φλάνδρας, και τους ομιλητές που θα μας παρουσιάσουν τις εργασίες. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Τσβέρ για τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις. Έχετε το λόγο, συνάδελφε Τσβέρ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επίσης ε, γιατί προκαλέσαμε ενδιαφέρον και ήρθαν αρκετοί στη σημερινή συνάντηση και σας ευχαριστώ επίσης ότι υπάρχει και σλοβενική διαρμηνία. Χαίρομαι γιατί μπόρεσα να προετοιμάσω την πρώτη αυτή έκθεση από κοινού με την κυρία Λομπάτσκα και άλλους συναδέλφους Έχω την εντύπωση ότι η έκθεση αυτή θα είναι ιδιαίτερο ωφέλιμη και για άλλες εκθέσεις, μέσω των οποίων θα αξιολογήσουμε την εφαρμογή του Erasmus+. Plus. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία αυτή σήμερα. Στηρίζω το Erasmus Plus. Γνωρίζουμε ότι το Erasmus Plus δημιουργήθηκε το 2014. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε και πάρα πολλά δεδομένα πάνω στα οποία να έδρασουμε την ανάλυση μας. Και φυσικά δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα. Παρότι όμως δεν έχουμε τα δεδομένα αυτά, στο τέλος του χρόνου οι πληροφορίες θα είναι αρκετές νομίζω, αφού υιοθετηθεί η έκθεσή μας ε, νομίζω ότι η έκθεσή μας έχει πολύ ενδιαφέρον. Ε, έχω έρθει σε επαφή με πολλούς εμπλεκομένους και θα συνεχίσω να το κάνω. Είχα πάρα πολλές διαβουλεύσεις. Όπως είπε και η πρόεδρος Κώστα, ήδη έχουν υπάρξει κάποιες σημαντικές μελέτες. Αυτές οι πρώτες μελέτες, αυτές οι πρώτες αξιολογήσεις νομίζω ότι μας δίνουν κάποιες ιδέες ε, στα πλαίσια της ε, ε, κρίσης μας γύρω από το Erasmus+. Έχοντας διαβάσει προσεκτικά λοιπόν αυτές τις μελέτες, μπορώ να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι από μεθοδολογικής επόψεως είναι ιδιαίτερως καλογραμμένες. Ως εκ τούτου τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν θα μπορούσαν να είναι έγκυρα. Επίσης θεωρώ ότι τα δικά μας συμπεράσματα που θα συμπεριλάβουμε ενώ στην δική μας έκθεση σαν Κοινοβούλιο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν συζητάμε τα θέματα εφαρμογής στο μέλλον. Το Νοέμβριο του 2015 διοργάνωσα μία συνάντηση σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση και τη μαθητεία. Οργανώσαμε επίσης και μία διάσκεψη για το Erasmus ε, Plus. Έχουμε και άλλες συναντήσεις προβλέψει, όχι μόνο τη σημερινή. Έχουμε επίσης ε, και τη δημόσια ακρόαση του ΕΛΚ για το Erasmus Plus ε, που θα ασχοληθεί με τον ρόλο τον οποίο παίζουν συνολικότερα οι νέοι στην Ευρώπη. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο ε, προηγήθηκε η πρώτη αντίστοιχη συνάντηση για τις τυπικές μορφές, παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης. Θα έχουμε επίσης ε, μία συνάντηση με ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ίσως τον κ. νομίζω ότι είχαμε την δυνατότητα λοιπόν να ανταλλάξουμε αρκετές πληροφορίες μέχρι τώρα, να συλλέξουμε επίσης αρκετές πληροφορίες Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του Erasmus Plus, βελτίωση ικανοτήτων, βελτίωση απασχολησιμότητας, προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος των κενών στις επαγγελματικέ γνώσεις. Το νέο πρόγραμμα προσπαθεί να τα απλοποιήσει τα πράγματα και να διασυνδέσει διαφορετικούς μεταξύ τους τομείς, έτσι ώστε όλοι να εμπλέκονται και να παίζουν τον ρόλο τους. Οι ασχολούμενοι με αυτά μας είπαν ότι υπάρχουν όμως προβλήματα, ότι τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσουν είναι περίπλοκα, οι σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δύσκολη και ότι υπάρχει έλλειψη χρημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της προσπαθεί να ξεπεράσει αυτά τα αρχικά προβλήματα στη λειτουργία του προγράμματος, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν είναι πλέον εφικτό να επιστρέψει κανείς στο παλαιό πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι κάποια προγράμματα πρέπει να συγκρατήσουν τα παλαιά τους ονόματα, όπως Comenius Grundvik ε, Λεωνάρντο Νταβίντσι ε, και τα λοιπά. Τα ονόματα αυτά πρέπει να παραμείνουν, είναι αναγνωρίσιμα. Έχουμε επίσης και τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, έχουμε τη στρατηγική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, έχουμε την γενικότερη στρατηγική για την νεότητα, ξέρουμε τους στόχους όλων αυτών των επιμέρους στρατηγικών Οφείλουμε όμως να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας και σε άλλους τομείς όπως οι μετανάστες. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε οι μετανάστες να μπορούν να συμμετέχουν στα κοινωνικά δρόμενα. 15 εθνικές αντιπροσωπείες συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Μέχρι σήμερα χρησιμοποίησαν το 100% των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων. Αυτό μας δείχνει ότι το πρόγραμμα λειτουργεί με επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Το πρόγραμμα αυτό βέβαια δεν είναι αυτόνομο, δεν είναι αυτάρκες, πρέπει να συνδεθεί με άλλους ευρύτερους τομείς όπως ε, η εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα, Υπάρχει ένα δίκτυο γύρω από το Erasmus το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς. Έχουμε τον συνδυασμό τομεακών αρμοδιοτήτων και γνώσεων. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, πολλαπλές μορφές δικτύωσης. Έχουμε εθελοντικές ενώσεις και υπηρεσίες κτλ εμείς μιλούσαμε για την τελευταία γενεά η οποία είχε προβλήματα απασχόλησης. Τώρα βλέπουμε ότι ο αριθμός των νέων που έχουν βρει δουλειά έχει κάπως αυξηθεί και σε ένα βαθμό υπεύθυνο σε εισαγωγικά γι' αυτό είναι και το Erasmus Plus. Τελειώνοντας λοιπόν θα πω ότι ήταν επιτυχές το Erasmus Plus. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για τις ε, πληροφορίες. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις εμπειρογνώμονές μας και να κάνουμε αυτή την πρώτη συζήτηση για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση που υπενθυμίζω ότι θα υποβληθεί τον Οκτώβριο. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο κύριε Βάχτερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω να μ' ακούτε, αλλιώς θα ουρλιάζω. Πέστε μου, σε 10 λεπτά ελπίζω θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης για την εφαρμογή των πρώτων ετών και τις πρώτες εμπειρίες ε, της εφαρμογής ε, του Erasmus ε, Plus. Όσον αφορά τις αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος, εσείς είστε ειδικοί σε θέματα παιδείας και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό εάν ε, δυσκολέψουν τα πράγματα και δεν ξέρετε πού βρισκόμαστε στις διαφάνειες, έχουμε εδώ τρία βήματα και θα προσπαθήσω να ακολουθήσω αυτά τα τρία βήματα. Θα σας κάνω πρώτα μια εισαγωγή και θα σας πω και δύο λόγια για τη μεθοδολογία. Στη συνέχεια θα σας πω τα βασικά μας ευρήματα σε μια ε, εικόνα και από εκεί και πέρα τα βασικά ευρήματα θα τα αναπτύξω λίγο περαιτέρω. η εισαγωγή και η μεθοδολογία. Ποιος έκανε αυτή τη μελέτη, η οργάνωση την οποία ευθύνω, ε, η Ένωση Ακαδημαϊκής Συνεργασίας και έγινε μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2016. Φρέσκο πράγμα. Ε, πέραν εμού ήταν η Μαρίγια Μίτιτς που είναι εδώ σήμερα και η Ειρήνα Φέρεντς επίσης. Ε, στόχος και πεδίο εφαρμογή προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε και να αναλύσουμε τις πρώτες εμπειρίες ε, με την εφαρμογή του Erasmus Plus και επικεντρωθήκαμε διότι αυτή ήταν και η εντολή που ε, μας έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για στις αποκεντρωμένες δράσεις και μόνο δράσεις οι οποίες κυρίως εφαρμόζονται από τις λεγόμενες εθνικές υπηρεσίες. Έγινε μια διαδικτυακή έρευνα για όλους αυτές τις υπηρεσίες ε, στην Ευρώπη, 61 τον αριθμό. Ε, λάβαμε απαντήσεις ε, παρεπιπτόντος με τον ένα με τον άλλο τρόπο από 40 εξ αυτών. με οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό και είχαμε και κάποιες συνεντεύξεις μέσω Skype. Περνάμε τώρα στην ευρύτερη εικόνα ρωτήσαμε πρώτα τι κατά την άποψή σας αποτελεί τα τέσσερα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτού του νέου προγράμματος και ποια είναι τα τέσσερα αρνητικά στοιχεία. Τα δύο τρίτα και πάνω των εθνικών υπηρεσιών θεώρησαν ότι η δυνατότητα ε, διατομιακής συνεργασίας ήταν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα τουλάχιστον η πλειοψηφία αυτό πιστεύει. Αλλά πρέπει να τονίσω ότι εδώ είναι δυνητικό το θέμα, διότι το πρόγραμμα όταν θα αναπτυχθεί περαιτέρω θα μας δείξει, όταν θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία, πόσο από αυτά τα πράγματα έχουν υλοποιηθεί. Δεύτερον, η αρχιτεκτονική δομή του προγράμματος που είναι εξορθολογημένη. Ε, ξέρετε, πλέον δεν βασίζεται ε, στο παλιό σύστημα. Πριν ήμασταν ε, επικεντρωμένοι σε συγκεκριμένου τομεί, παραδείγματο χάρη στην εκπαίδευση, αλλά τώρα έχουμε μια λογική δραστηριότητα και από εκεί έχουμε τι βασικέ μα δράσει απλοποιημένη οικονομική διαχείριση, κυρίως υπό τη μορφή κόστους αναμονάδα και εδώ έχουμε και πάλι δυνατότητες για μεγαλύτερη επιρροή υπό την έννοια ε, των στόχων πολιτικής που έχει καθορίσει το πρόγραμμα ε, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε τα μειονεκτήματα. Περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτό είναι εμφυβισμός περιορισμένη λειτουργικότητα εργαλείων πληροφορικής ε, και του βασικού αριθμού. Έχουμε πάρα πολλά και πολύ κακά εργαλεία πληροφορικής και αυτή ήταν η βασική ε, ε, αρνητική πτυχή περίπλοκα διοικητικά θέματα και γραφειοκρατία, αυτή ήταν η συνέχεια. Το 75% είπε ότι έχουν γίνει αξιολογήσεις προγράμματος από τη δεκαετία του 80 και πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά την απλούστευση, κανείς ποτέ δεν είναι ικανοποιημένο. Αυτό δεν χρειάζεται λοιπόν να το δραματοποιούμε. Ε, προτίμηση για... Ε, προγράμματα μεγαλύτερης κλίμακας ε, σημαίνει ότι είναι δυσαρεστημένοι αυτοί που κάνουν αιτήσει για μικρότερα προγράμματα. Παραδείγματος χάρη στην ε, τομέα των νέων που θεωρούν ότι προτιμούν μεγαλύτερα προγράμματα ε, και ότι κυρίως οι νέοι που κάνουν αιτήσει δεν θα έχουν ισότιμη μεταχείριση. Και εναρμόνιση ε, ανατομέα, αυτή έχει υπερβεί λίγο κάποια όρια και αυτό εξέφεσαν κάποιο αρνητικό στοιχείο. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες. Δυνατότητες για διατομιακή συνεργασία. Ρωτήσαμε πώς πηγαίνει αυτό το πράγμα. Αυτή ήταν μία από τις μεγάλες προσδοκίες του νέου προγράμματος. Είναι πολύ νωρί για να απαντήσουμε βάσει τα ε, ασφαλών εμπειρικών ε, στοιχείων, αλλά όταν ρωτήσουμε όσον αφορά τι προσδοκίε και τι πρώτε εμπειρίε, δεν βλέπουμε τόσε μεγάλες αλλαγέ σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. 1,65% θεωρεί ότι υπάρχει μια μέτρια αύξηση ε, διατομιακή ε, συνεργασίας. Ένα 8,6% θεωρεί ότι είναι ουσιαστική άξιση και ένα 25% περίπου θεωρεί ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες αύξησης, αλλά δεν ε, γίνεται γρήγορα αυτή η αύξηση, δεν εκτοξεύεται εν μία νυχτή. Ε, η έλλειψη σαφήνειας ε, είναι κάτι για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν κάποιες υπηρεσίες ε, για το τι ακριβώς είναι η διατομιακή συνεργασία και ζητούσαν ορισμούς από αυτόν. Η σύστασή μας είναι η διατομιακή συνεργασία πρέπει να εκτελεστεί, να υλοποιηθεί, να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί στην πράξη. Επόμενη. εξορθολογημός των κανόνων του προγράμματος σε κάθε τομέα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος και έγιναν ε, δύσκολες συζητήσεις και στο παρελθόν πριν εφαρμοστεί το πρόγραμμα για το κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα ή όχι. Κατά την άποψη των υπηρεσιών, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία αλλαγή για τον τελικό χρήστη, για τους φοιτητέ, το προσωπικό τους νέους και ε, αυτούς που υποβάλλουν αιτήσει, καθώς επίσης και για το ESEA, αν και εγώ αναρωτιέμαι πώς το ξέρουν αυτό, γιατί δεν συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μια αλλαγή προς το χειρότερο θεωρούν για τον εαυτό τους. Ε, έχουν περισσότερη δουλειά, τους επιβαρύνει περαιτέρω. Αλλαγή προς το καλύτερο θεωρούν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω ε, αν αυτό είναι επειδή πιστεύουν πάντα ότι οι άλλοι ζουν καλύτερα και είναι πιο εύκολα τα πράγματα για αυτούς, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω εικασίες εδώ. Τώρα, για το τομέα της νεολαίας, τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο θετικά. Ε, εδώ έχω μια παράθεση για τους νέους, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εναρμόνιση, 40% των ετούντων χάθηκαν στον πρώτο χρόνο. Η σύστασή μας είναι να μην υπάρχει άλλη εναρμόνιση, Καλό είναι το γεγονός ότι υπήρξε εναρμόνιση, αλλά πλέον πρέπει να ε, παγιωθούν κάποια πράγματα, ε, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ε, καλά στοιχεία. Η οικονομική διαχείριση πάντα είναι σοβαρό θέμα σε όλα τα προγράμματα ε, από την αρχή των προγραμμάτων τους ε, ε, και το αεράσμους ή το κόμετ που είχαμε στη δεκαετία του 80. Εδώ είχαμε ένα κόστος αναμονάδα και συνολικά ποσά τα οποία διευκόλυναν την οικονομική διαχείριση θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους δικαιούχους του προγράμματος και ένα 54,3% των εθνικών υπηρεσιών θεωρεί ότι οι δικαιούχοι πλέον διευκολύνονται περισσότερο. Ένα 20% θεωρεί ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα και μόνο ένα 25% θεωρεί ότι η δουλειά τους είναι πιο επαχθής. Περισσότερο από αυτούς που ε, δικαιούνται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δηλαδή. Ε, για τις υπηρεσίες η αλλαγή δεν ήταν τόσο εμφανής. Ε, ένα ε, 44% πιστεύει ότι διευκολύνθηκε η δουλειά του. Ένα 16,7% θεωρεί ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και περίπου ένα 40% πιστεύει ότι έχει γίνει πιο επαχθής. Ε, νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχει σαφής ε, τάση, είναι λίγο ανάμεικτα τα πράγματα, αλλά ε, υπό την έννοια της διευκόλυνσης της οικονομικής διαχείρισης ε, πιστεύουν ότι επιβαρύνονται από γραφειοκρατία λού, υπερβολικούς ελέγχους, υπάρχει το θέμα το, της πληροφορικής, προβλήματα με τις Οδηγίε κλπ. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση. Ε, το Εράσμους χρηματοδοτείται καλά ή χρηματοδοτείται παρκώς. Ένα 50% θεωρεί ότι χρηματοδοτείται παρκώς. Οι υπόλοιποι είναι κάτι σαν το Brexit. Σχεδόν το ίδιο ποσοστό θεωρεί ότι δεν χρηματοδοτείται παρκώς. Δεν υπάρχει καμία υπηρεσία παρεπιπτόντω που να θεωρεί ότι ε, χρηματοδοτείται υπερβολικά αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει. Όσον αφορά τις βασικές δράσεις και τους διάφορους τομείς, η εικόνα γίνεται λίγο πιο θολή. Ε, το KA2 θεωρήθηκε ότι δεν χρηματοδοτείται αρκετά ε, για, από τα 4 πέμπτα των ε, όσων απάντησαν. Το KA3 θεωρείται ότι ε, χρηματοδοτείται επαρκώς, ε, κυρίως από την πλειοψηφία των υπηρεσιών, περίπου τα 2 τρίτα. και το KA της κινητικότητας είναι κάπου ενδιάμεσα. Ανατομέα, η εκπαίδευση των ενηλίκων υποχρηματοδοτείται, ε, θεωρούν οι περισσότεροι, ένα 81% και στη συνέχεια οι νέοι και η σχολική εκπαίδευση. Η επαγγελματική ε, κατάρτιση είναι ο μόνος τομέας, και αυτό με εξέπληξε, όπου η πλειοψηφία θεωρούν ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Τα καταποκοπήν ποσά ε, θεωρήθηκαν ε, πολύ καλή λύση, αλλά το θέμα είναι κατά πόσον επαρκούν. Ε, υπήρχαν αρκετές επικρίσεις, όχι δεν επαρκούν και καλύπτουν πολύ λιγότερα από όσα κάλυπταν στα προηγούμενα προγράμματα όταν δεν υπήρχε απαραίτητα ένα καταποκοπήν ποσήν αλλά υπήρχε και ένα επίπεδο χρηματοδότησης. Η σύστασή μας είναι η οποία δεν βασίζεται στην πραγματικότητα σε καμία από αυτές τις παρατηρήσεις που σας ανέφερα προηγουμένως, ε, διότι ορισμένες φορές μας είπαν ότι τους απομένουν και κονδύλια για ένα τμήμα του προγράμματος, ενώ χρειάζονται κονδύλια για άλλο τμήμα του προγράμματος, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν μεταφορά των κονδυλίων λόγω περίπλοκων κανόνων προπολογισμού που δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι ετούντες και οι δικαιούχοι του προγράμματος. Το πρόγραμμα θέλει να προσελκύσει νέες μορφές οργανισμών. Η μεγαλύτερη αντιληπτή αύξηση νέων ε, είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, περίπου ένα 50%, δημόσιοι φορείς επίσης με 45% και επιχειρήσεις ε, κάτι λιγότερο του 40%. Το μεγαλύτερο μερίδιο των υπηρεσιών όμως θεωρεί ότι η συμμετοχή αυτών δεν έχει ούτε αυξηθεί ούτε μειωθεί ε, είναι σχεδόν αντίστοιχο το μερίδιο, επομένως δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και το Erasmus Plus, όπως σας είπα και προηγουμένως, θεωρείται ότι ευνοεί μεγάλα προγράμματα και δεν ευνοεί μικρότερες οργανώσεις που δεν είναι τόσο καλά εξοπλισμένοι στον τομέα των νέων, για παράδειγμα, αλλά όχι μόνο εκεί. Υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα σε κάποιες δράσεις, για παράδειγμα στην KA2, βασική δράση 2 και κυρίως ε, τις ε, στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις, όπου σε κάποιες περιπτώσεις τα ποσοστά αποδοχής είναι κάτω του 10%. Και αυτό φυσικά μπορεί να αποτελέσει και κίνδυνο για το πρόγραμμα, διότι ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον ότι έχουν μια σοβαρή ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν. Τελειώνω σχεδόν κόκκινο στόχο, αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο, να δούμε ε, και αυτέ τι κατηγορίες, άτομα ε, με, ε, από ευάλωτο παρελθόν ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Ε, τα άτομα με ειδικέ ανάγκε εδώ δεν έχουμε μεγάλε αλλαγέ σε σχέση με τα προηγούμενα στο παρελθόν προγράμματα ε, και άτομα από πιο ευάλωτο παρελθόν η, μια μικρή πλειοψηφία θεωρεί ότι το Erasmus Plus είναι δυνητικά καλύτερα εξοπλισμένο να αντιμετωπίσει τις ανάγκες από ό,τι τα προηγούμενα προγράμματα. Η η πρότασή μας είναι να αφήσουμε περιθώριο και για αιτήσει από ε, προγράμματα ή από ε, περιπτώσεις όπου έχουμε μικρότερους ε, ετούντες. Τώρα, συνεργασία μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών και αυτών που οποίων εφαρμόζουν το πρόγραμμα. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίπου η μισή από όλες τις υπηρεσίες είτε είναι ικανοποιημένη είτε πολύ ικανοποιημένη με τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα 30% δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένη και περίπου μόνο το 1 πέμπτο είναι δυσαρεστημένο ή πολύ δυσαρεστημένο. Το μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης είναι με αυτό το οποίο αποκαλούμε το πλήρες ε, χαρτοφυλάκιο, το υπηρεσίε μάλλον πλήρους χαρτοφυλακίου, δηλαδή οι υπηρεσίε οι οποίες είναι αρμόδια για όλα τα τμήματα του προγράμματος. Αν είχαμε θέσει αυτή την ερώτηση ε, πριν από ένα χρόνο η απάντηση θα ήταν πολύ πιο αρνητική. Έχει υπάρξει ε, πρόοδος παρά το γεγονός ότι η αρχή ήταν κάπως δύσκολη και έγιναν προσπάθειες από όλους τους για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Τώρα, συνεργασία με τον εκτελεστικό φορέα. Ε, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος τώρα με τη διατύπωση εδώ. Ε, τελειώνω σε ένα λεπτάκι. Υπάρχει σχεδόν μηδενική συνεργασία. Αυτό πρέπει να αναφέρεται εδώ, διότι οι δύο οργανισμοί ε, αφορούν τελείως διαφορετικό τμήμα του προγράμματος, αλλά υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία, κυρίως σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών, γιατί και οι δύο ενημερώνουν για τα τμήματα του προγράμματος Erasmus Plus που δεν είναι αρμόδιοι Επομένως, ε, μια πιο επίσημη, πιο συστηματική συνεργασία με την, ε, υπηρεσία, ε, την εκτελεστική υπηρεσία. Θα παρακάμψω τα εργαλεία πληροφορικής, τα έχετε ακούσει 100 φορές, είναι μια καταστροφή την οποία ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να μετριάσουμε, αλλά γίνονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Η σύσταση είναι να μην γίνουν περισσότερα, αλλά να έχουμε λιγότερα και καλύτερα εργαλεία πληροφορικής. Και μια τελευταία παρατήρηση. Διαπιστώνουμε ότι το πρόγραμμα έχει ε, τύχει προώθηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους ενδιαφερομένους και από όλους. Σε κάποιο βαθμό αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και τεράστια απογοήτευση, διότι αν εξετάσετε κάποιες δράσεις, όπου η κάθε χώρα έχει ελάχιστες υποτροφίες, για παράδειγμα, για την ε, ε, κινητικότητα σε μη ευρωπαϊκές χώρες, ε, τότε μπορεί να μην έχουμε σωστά αποτελέσματα. Επομένως, προτείνουμε να επικεντρωθούμε στα τμήματα του προγράμματος που δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς. Να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και να σας δώσω και μία τελευταία σύσταση που μας διαβίβασαν οι υπηρεσίες. Όλα αυτά ήταν πολύ καλά, όλη η μεταρρύθμιση ήταν καλή, αλλά αυτή τη στιγμή φτάνει πια, όχι άλλες αλλαγές απλώς για να αλλάζουμε τα πράγματα. Ας προσπαθήσουμε να δούμε τι έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you so much. Very, very interesting this study. ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες της παρουσιάσεις και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κετούνεν. 10 λεπτά. Από το EPRS. Κυρίες και κύριοι, και τον ονομάζομαι. Και είμαι από την, ε, το Πανεπιστήμιο του Τουρκού. Και ρόλος μου είναι να αξιολογήσω το, την, ε, το εργαλείο για την αξιολόγηση του, της πρόοδου του Εράσμου. Το πλαίσιο λοιπόν ε, αξιολόγησης είναι αρκετά απλό και βασίζεται στο γεγονός ότι στα project χρειάζομαστε δύο πράγματα. Καταρχάς, χρειαζόμαστε χρηματοδότηση και κατά δεύτερον, ικανότητες και προσόντα. Και σε συνέχεια αυτών μπορούμε να περιμένουμε κάποιες ενέργειες και δράσεις σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες, ανάλογα τον κλάδο και την ανάπτυξη δυναμικού και αναμένουμε και κάποιον αντίκτυπο βάσει των δράσεων αυτών ασφαλώς. Ας αναλύσουμε λοιπόν την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus Plus από την πλευρά αυτή, από την οπτική γωνία αυτή, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τις ικανότητες αυτές. Γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά για το πρόγραμμα. Να πω από πλευρά αντικτύπου ότι ο εξωτερικό αντικτύπος των ενεργειών των δράσεων αυτών μπορεί να αυξηθεί θέτοντας προϋπόθεση και απέτηση να υπάρχουν πιο πολλές οργανώσεις και ενδιάμεσες οργανώσεις, για παράδειγμα επιχειρήσεις και άλλες οργανώσεις πελατών. Και αυτό γιατί η καινοτομία αποτελεί ένα βασικό στόχο του προγράμματος. Και η καινοτομία μπορεί να βελτιωθεί από τις απαιτήσει που περιλαμβάνονται στον οδηγό του Erasmus Plus σε ό,τι αφορά την προετοιμασία και των προτάσεων προγραμμάτων και έργων, εφόσον η καινοτομία περιλαμβάνεται εξ αρχή. Και οι καινοτομίε λοιπόν είναι απλά ιδέε οι οποίε έχουν εφαρμοστεί σε επιχειρήσει και το δημόσιο κλάδο. Από πλευρά χρηματοδότηση, δε, θα ήθελα να πω το εξή. Αν υπάρχουν σημαντικοί πολιτικοί στόχοι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδική, ειδικές δαπάνε, ειδική πόρη για να χρηματοδοτηθούν αυτοί οι, οι στόχοι. Για παράδειγμα, ένας από αυτού είναι και η πολυγλωσία. Ενδεχομένω να υπάρχουν και άλλοι, άλλες πολιτικά σημαντικέ δραστηριότητε. Και τα προγράμματα αυτά, τα έργα αυτά, περιλαμβάνουν και πάρα πολύ χαρτούρα. Αυτό θα πρέπει να περιοριστεί προκειμένου η χρηματοδότηση να έχει ως στόχο τα πιο σημαντικά στοιχεία των προγραμμάτων. Τώρα, οι κανονισμοί για την ε, την ισότητα μεταξύ των ατόμων στα project ε, δεν έχει πολύ νόημα. Γιατί για τις ε, άλλες οργανώσεις τέτοια προγράμματα δεν είναι και ιδιαίτερα υποφελή. Αν λοιπόν και άρα χρησιμοποιούνται κατά βάση χαμηλόμισθοι σε αυτά τα project. Αντί να χρησιμοποιούνται υψηλόβαθμα στελέχη ε, και ακαδημαϊκοί επίσης υψηλόβαθμοι. Άρα δεν βοηθάει αυτή η αρχή για την ίση αμοιβή θα πρέπει να περιλαμβάνονται περιγραφές σε ό,τι αφορά τις δομές που χρησιμοποιούνται στα project, προκειμένου να επιτευχθεί το ευκταίο αποτέλεσμα και οι δραστηριότητε θα πρέπει να είναι evidence-based, βάσει συγκεκριμένων τεκμηρίων, προκειμένου να είμαστε, ε, να περιμένουμε και κάποιο αντίκτυπο από τις δραστηριότητε και θα πρέπει να βασίζονται στην ιδέα που θα ισχύει και για τις επιχειρήσεις και για τις άλλες οργανώσεις ε, καταναλωτών. Και τέλος και τα θέματα βιωσιμότητας και διάδοσης των ε, project θα πρέπει να εξασφαλίζονται μέσω της χρήσης υφιστάμενων και καινούριων, μόνιμων δομών, τα, οι οποίες θα υπάρχουν και μετά την ε, παρέλευση και τη λήξη των project. Προκειμένου λοιπόν να συνεχίσει η διάσταση αυτή της βιωσιμότητας του έργου και μετά την περάτωση του έργου. Οι ικανότητε τώρα και τα προσόντα. Θα ήθελα να πω το εξή εδώ. Το πρόγραμμα Erasmus Plus θα πρέπει να κάνει μία σαφή αναφορά στα ευρωπαϊκά εργαλεία για τη διαφάνεια και την αναγνώριση και το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Πολλά project δεν χρησιμοποιούν το καλύτερο το προσωπικό. Και θα πρέπει να υπάρχουν άτομα τα οποία θα έχουν και μεταπτυχιακές σπουδέ και διδακτορικό στο αντικείμενο των project. Και τα κατήρια θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και σχετική εμπειρία, προηγούμενες δημοσιεύσεις για τα θέματα αυτά και μια διεθνή εμπειρία. Μίλησα δε και με πολλούς εμπειρογνώμονες από άλλε χώρε. Και τα αποτελέσματα στα οποία καταλήξαμε είναι τα εξή. Συνομιλήσαμε και κάναμε συνεντεύξεις και με τα στελέχη των ε, project και με πολλούς πολλούς εμπειρογνώμονες. Και βλέπετε λοιπόν ποιες είναι οι συστάσεις βάσει των συνεντεύξεων αυτών. Το ευθέω λοιπόν αποτέλεσμα των project μπορεί να επιτευχθεί πιο άνετα, δίνοντας πιο πολλούς πόρους στα σημεία α, κλειδί των project, προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί προγραμματικοί στόχοι. Κάποια στιγμή κάποιος είχε πει ότι περίπου 40% των οικονομικών πόρων χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των project αυτών. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ε, σκόπιμο. Θα πρέπει η ουσία να χρηματοδοτείται και όχι τα γύρω-γύρω. Και επίσης ε, να μην έχουμε περιττή γραφειοκρατία και χαρτούρα μεταξύ των ε, αρμόδιων οργάνων. Και επίση χρειάζονται ένα έλεγχο των εθνικών χρηματοδοτήσεων, μεγαλύτερη αυτονομία και πιο απλοί κανόνε. Και πιστεύουμε ότι η ποιότητα των project μπορούν, μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω στη φάση της προετοιμασίας των έργων, γιατί συνήθως δεν υπάρχει χρόνος για την σωστή προετοιμασία και γενικώ υπάρχουν πολλές ε, προτάσεις για project οι οποίες ε, είναι στη φάση της προετοιμασίας. Έτσι, αν είχαμε πιο πολύ χρόνο, θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε και πιο πολύ χρόνο για την προετοιμασία της πρότασης και έτσι να βελτιωθεί και η ίδια η ποιότητα του project. Η μεγαλύτερη λοιπόν πρόκληση είναι θα μπορούσε μάλλον να αντιμετωπιστεί με μία πλατφόρμα, διαδικτυακή πλατφόρμα, προκειμένου να απλοποιηθεί η χρήση των εργαλείων εφαρμογής και να απλοποιηθεί η διαχείριση, η εφαρμογή, ο έλεγχος κτλ. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια μεγάλη πρόκληση για να μειωθεί πια η περιττή πραγματικά σε ένα βαθμό γραφειοκρατία και να εστιαθούμε πιο πολύ στην ε, ουσία των προγραμμάτων. Αυτή είναι λοιπόν ε, η μεγάλη πρόκληση και έτσι ολοκληρώνω την παρουσίασή μου και σας ευχαριστώ Σας Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος για τις πολύ χρήσιμες αυτές τις στάσεις. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βίκ για 7 λεπτά για το λόγο. Yes, thank you, Chair. Uh, my name is Hans Vika. I am the head of Jugendführung. Λέγομαι Βίκε. For Youth in Action. And we are one of four national agencies in Germany. Μας μία από τις τέσσερις εθνικές υπηρεσίες στην Γερμανία που ασχολούμεθα με τέτοια θέματα. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, δεν είναι πρόβλημα το ότι είμαστε τέσσερις. έχουμε αρκετά καλή συνεργασία λοιπόν. Θα πρέπει επίσης να πούμε και θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσβέρ για τις εμπειρίες τις οποίες έχει καταλήξει ότι το πρόβλημα μέχρι τώρα είναι σχετικά επιτυχές. Αν δει κανεί τους αριθμούς ήδη από το 2016, βλέπουμε ότι έχουμε εξίσου μεγάλο αριθμό υποψηφιωτήτων με το 2014. Έχουμε δαπανίσει το σύνολο των διαθέσιμων πιστώσεων. Τα νέα φορμάτα, τα οποία είναι στη διάθεσή μας έχουν αρχίσει να λειτουργούν καλά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν ε, τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας όπως λένε, αλλά παρόλα αυτά βελτιώνουμε πάρα πολύ τις εμπειρίες των νέων. Στα πλαίσια της διαχείρισης κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στους ε, πραγματικούς πρωταγωνιστές, δηλαδή τους νέους. Υπάρχει όμως ο χώρος προς βελτίωση και αυτό δεν εκπλήσει είναι ένα νέο πρόγραμμα συνεργαζόμαστε σωστά και με τα προγράμματα τα οποία ανήκουν στον κύκλο της διαβίου κατάρτισης σαν παράδειγμα όπου και εκεί θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό κεφάλαιο για τους νέους. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη σημασία που έχει αυτή η κοινωνική κατηγορία. Δεν είναι μόνο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμείς είμαστε ένα κομμάτι του ευρύτερου στρατηγικού πλαισίου για την νεότητα. Είναι σημαντικό αυτό και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί συγκεκριμένους περιορισμούς στα πλαίσια των δυνατοτήτων, α, περαιτέρω μάλλον δυνατοτήτων εναρμόνισης. Έχει ήδη υποθεί ότι σε ορισμένα επίπεδα η εναρμόνιση θα πρέπει να σταματήσει κατά κάποιο τρόπο. Αυτή είναι μια εντύπωση που διαμορφώθηκε. Βλέπουμε όμως ότι σε κάθε ένα τομέα ξεχωριστά και δεν μιλάμε μόνο για το Youth in Action, αν θέλουμε πραγματικά να αποτυπώσουμε το ίχνος μας στον τομέα αυτό των σπουδών, ε, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες τομιακές, τομιακές συνεργασίες. Έτσι θα καταστήσουμε τη ζωή των νέων ευκολότερη, την εκπαιδευτική τους εμπειρία και θα έχουμε και μία στρατηγική εφαρμογή των ρυθμίσεων η οποία θα είναι πιο αποτελεσματική. Τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν κάτι έχουμε πετύχει. Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα θα έλεγε σημαντικές. Έτσι θα πετύχουμε τους βασικούς στόχους του προγράμματος Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν και από τις Εθνικές Υπηρεσίες Εράσμους και από τις Κοινοτικές Υπηρεσίες. Για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να πούμε και ίσως να μην το γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή για το Youth in Action, 10%. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και αυτός ο περιορισμός αν θέλετε στην χρηματοδοτική ευελιξία δίδει κάποιες εγγυήσει για την σωστή χρήση του προϋπολογισμού για τους νέους και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι με το 10% του προϋπολογισμού έχουμε το 25% των συμμετοχών έχουμε αν θέλετε ένα υψηλότατο επίπεδο συμμετοχής και ένα υψηλότατο αριθμό δραστήριων οργανώσεων. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για αυτά τα οποία κάνει το Youth in Action εφόσον υπάρξει κάποτε και ελπίζουμε να έρθει το 2017 ή το 2018 μια τέτοια αύξηση, δεν θα έχουμε καμιά τέτοια δυσκολία για τη χρήση του προϋπολογισμού, θα υπάρξουν αντίθετα περαιτέρω χρηματοδοτικές ανάγκες. Αυτά λοιπόν για το Youth in Action. Τώρα για τη διατομεακή συνεργασία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τεράστια, θα έλεγα τεράστιο πεδίο συνεργασίας. Δεν έχουμε πετύχει ακόμα ε, την ολοκλήρωση της διατομεακής αυτής συνεργασίας. Αυτό δεν γίνεται γιατί δεν το επιθυμούμε ή γιατί δεν το επιθυμούν οι συμμετέχοντες. Αυτό οφείλεται γιατί υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες. Για να το πετύχουμε θα πρέπει να έχουμε τα σωστά μέτρα, τα σωστά έντυπα και έγγραφα, την σωστή υποστήριξη. Θα πρέπει ίσως να υπάρχουν και συγκεκριμένες διαφορετικού τύπου επιμέρους δράσεις για αυτό που θα ονομάζουμε από εδώ και πέρα διατομιακή συνεργασία. Erasmus Plus. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι περαιτέρω γραφειοκρατικό άχθος. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Είναι ιδιαίτερος περίπλοκο το πρόγραμμα. Η δυσκολία αυτή είναι σαφής και γι' αυτό και γίνονται προσπάθειες και πολλές από αυτές είναι επιτυχείς έτσι ώστε να μειωθεί αυτό το γραφειοκρατικό άχθος. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε να προσπαθήσουμε να το μειώσουμε και για αυτούς που καταφέτουν αιτήσει και για τις διοικήσεις σε εθνικό επίπεδο. Να υπογραμμίσω επίσης ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές υπηρεσίες είναι κάτι το επιτυχές και στο Youth in Action και στο συνολικότερο Erasmus Plus. Έχουμε κοινέ στρατιστικές, στρατηγικές, συγγνώμη, έχουμε κοινά μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε και αυτό είναι μια καλή εγγύηση θα έλεγα για να καταλήγουμε στο τέλος με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η τυποποίηση είναι ένας τρόπος για να το πετύχουμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι η σωστή στενή συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές υπηρεσίες και στενή συνεργασία των εθνικών υπηρεσιών με την κοινωνία των πολιτών. Όλα αυτά στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής διάστασης. Αυτή λοιπόν η ευρωπαϊκή συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές υπηρεσίες, τα εθνικά γραφεία Erasmus Plus θα πρέπει περαιτέρω να ενισχυθεί αυτό για μένα είναι ένα θα έλεγα από τα στοιχεία που θα εγγυηθεί την θερμή υποστήριξη του προγράμματος από το κοινό. Ένα πρόγραμμα λοιπόν το οποίο είναι κοντά στον τελικό χρήστη, ένα πρόγραμμα σημαντικό και για το εθνικό επίπεδο, ένα πρόγραμμα και σημαντικό επίσης για το ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να διατηρηθεί λοιπόν ο αποκεντρωμένος εν μέρη χαρακτήρας του προγράμματος, από την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες μικιό ευρωπαϊκές που ζητούν να ληφθούν επιμέρους μέτρα, μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να, αντιμετωπίζουν προβλήματα σε συγκεντρωτικό επίπεδο, για να μην πω σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή στις Βρυξέλλες σεβόμενοι όπως πάντα τον αποκεντρικό, το μη συγκεντρωτικό χαρακτήρα του προγράμματος. Λοιπόν, σε μία από τις επιμέρους μελέτες λέγεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει τους τρόπους ε, αξιολόγησης ενδιάμεση σημεί των διαδικασιών του Erasmus Plus. Και αυτή είναι η σωστή πορεία ε, και για το επιμέρους πρόγραμμα με το οποίο ασχολούμαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Τράτσερτ. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να δω την αλλαγή προς το χειρότερο, αν κατάλαβα καλά από την ε, μελέτη της ε, ε, ΑΚΑ ε, έχει αλλάξει προς το χειρότερο κατάσταση για τις υπηρεσίες. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω μια μαρτυρία για το πώς εμείς ως υπηρεσία που ασχολείται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση εδώ στη Φλάνδρα αντιμετωπίσαμε ένα νέο πρόγραμμα και τι συνέπειες υπήρχαν για την εσωτερική μας οργάνωση. Καταρχάς, για δύο χρόνια ε, είχαμε το θέμα αυτό, το 2014 και το 2015, διότι δεν υπήρχε μετάβαση και ένα μεγάλο κενό μεταξύ του Erasmus ε, ε, Plus και του LLP. Έπρεπε να έχουμε τις τελευταίες εκθέσεις του LLP ε, που να συνδυάσουμε, να προωθήσουμε, να εξηγήσουμε και να δώσουμε συμβουλές για ένα νέο σχεδιασμό προγράμματος. Δεδομένου του γεγονότος ότι σε ένα πρόγραμμα διαβούη μάθησης με ε, διαφορετικές δράσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ήταν εύκολα τα πράγματα για τη διεθνή υπηρεσία. Είχαμε τέσσερις κλάδους, ο καθένας είχε τον κύκλο τους, του κανόνες του και κάναμε τα πάντα, από την ενημέρωση μέχρι την τελική έκθεση. Το 2014 και 2015 ήταν πολύ δύσκολο, διότι έπρεπε να γίνει μια εσωτερική αλλαγή από μια δομή που έκανε προσαρμογή για τη διαβίου και ταυτόχρονα μια άλλη δομή για να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα Erasmus+. Μάθαμε στην πράξη. Ε, το ίδιο έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι εθνικές υπηρεσίες ε, στον τομέα και είναι μια απλούστευση του προγράμματος, αλλά προσπαθήσαμε να ε, ερμηνεύσουμε και να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Από την άλλη, ενοιολογικά, με την εισαγωγή των αποκεντρωμένων στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και τις αλλαγές ε, για την ε, για την παιδεία είχαμε μεγάλες αλλαγές όχι μόνο για τις υπηρεσίες αλλά και για τον όλο κλάδο. Τώρα όλοι είμαστε υπέρ του Erasmus Plus, παρά το γεγονός ότι ήταν δύσκολη η προσαρμογή. Τώρα, για μας ω υπηρεσία, ε, τίθεται το ερώτημα τι προφίλ, τι πόρους, ε, τι ε, αρμοδιότητες χρειαζόμαστε ω Εθνική Υπηρεσία για να διαχειριστούμε αυτά τα προγράμματα. Διότι είναι διαφορετικό το πρόγραμμα, οι προσδοκίε είναι ε, διαφορετικές. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής ε, στο διαβίου μάθησε ε, έκανε κυρίως διαχειριστικά πράγματα, ενώ σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα και να, αφορά, να ασχολείται και με το περιεχόμενο του προγράμματος. Υπάρχουν νέες προσδοκίες όσον αφορά τις συνέπειες, ε, τη δημοσιοποίηση, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πόρους και αρμοδιότητες που δεν έχουμε σε αυτό το βαθμό και δεν είχαμε τουλάχιστον στη διάρκεια του προγράμματος. Είναι περίπλοκο αυτό και στην αρχή υπήρχαν πολύ μεγάλες προσδοκίες, υπήρχε και μια κάποια απογοήτευση και όπως είπε και ο συνάδελφος αλλάζουν όμως τα πράγματα πλέον. ένα από τα πρώτα στοιχεία που διαπιστώσαμε είναι ε, για ποιο λόγο να κάνει ένας οργανισμός έτσι για το Erasmus Plus. Και συχνά αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε αν το κάνουν για τα χρήματα ή για την διεθνή τους εικόνα. Κάθε χρόνο λαμβάνω τηλεφωνήματο κυρίως από ανώτατα εκπαιδευτικά ε, ιδρύματα, που με ρωτούν ε, ποιο είναι το μέγιστο ποσό για το οποίο μπορώ να κάνω αίτηση. Τα, τις αιτήσει μετά βλέπουμε ότι κάνουν έτσι για το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Ε, η ανώτατη εκπαίδευση βέβαια έχει κάποιες συγκεκριμένε ε, ε, δυνατότητες, αλλά στη σχολική εκπαίδευση ή σε επαγγελματικές σχολές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για τα κατάλληλα προγράμματα. Το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα δεν είναι καλό για ένα σχολείο και το να καταρτήσεις μία αίτηση, αν δεν έχεις κατάλληλο υπόβαθρο, δεν είναι πολύ καλό για σένα. Και φυσικά ε, οι εθνικές υπηρεσίες είχαν προβλήματα με τα προγράμματα πληροφορικής. Δεν θα σας πω τώρα τα της πληροφορικής, αλλά δυσκολευτήκαμε. Από την άλλη, Είχα το πλεονέκτημα ότι εγώ είμαι πελάτης ε, στη διαβίου μάθηση και διευθυντής ε, στο Erasmus Plus, επομένως μπορούσα να αλλάξω εστίαση όταν ξεκίνησα ως διευθυντής ε, του προγράμματος Erasmus Plus και ένα από τα βασικά οράματα, όχι δικό μου όραμα, αλλά από τις βαθικές οδηγίες που μου δώσανε ήταν κατευθυντήρες γραμμές από την Επιτροπή του Erasmus Plus για το τι ακριβώς κάνει μια εθνική υπηρεσία, τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία και έχουμε μια φράση εδώ από το 2014, ε, θεωρούν ότι είμαστε ε, άτομα που προωθούν το Erasmus Plus στην, ε, στην περιοχή μας. Είμαστε διαμεσολαβητές. Και να σας ε, καθησυχάσω και να σας διαβεβαιώσω ότι πολλοί από τους συναδέλφους έκαναν τις ίδιες συζητήσεις. Πώς μπορούμε να οργανωθούμε σε αυτή τη δομή του προγράμματος. Πρέπει εσωτερικά να υπάρχει απόφαση μεταξύ δράσης 1 και δράσης 2. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε την προσέγγιση ανατομέα. Ε, πρέπει να έχουμε ε, ταυτόχρονα και περιεχόμενο και διαχείριση. Είναι πολλές ερωτήσεις που έθεσαν και οι συνάδελφοι. Και όλα αυτά φυσικά πρέπει να τα μεταφράσουμε σε εκπαιδευτικά και προγράμματα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στο δικό σας το πεδίο. Παραδείγματο χάρη, επαγγελματική εκπαίδευση στη Φλάνδρα. Υπάρχουν σχολέ που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με γενική παιδεία. Ένα σχολείο λοιπόν που περιλαμβάνει και τι δύο μορφέ εκπαίδευση μπορεί να κάνει αίτηση και για τη σχολική εκπαίδευση και για την επαγγελματική εκπαίδευση. Επομένω είναι δύσκολη συζήτηση. Αυτό φυσικά οδήγησε και στο ερώτημα γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Τι φιλοδοξία έχουμε ως Εθνική Υπηρεσία, τι προσδοκίες υπάρχουν και ε, κυρίως τι πρόταση κάνουμε για να προσπαθούμε να προωθήσουμε. Ε, τους καλέσαμε για ένα φόρουμ ενδιαφερομένων και προς έκπληξή μας πάνω από 200 σχολεία και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ε, παρευρέθησαν. Στην αρχή περίμενα ότι θα διαμαρτυρηθούν για το Erasmus Plus, αλλά σύντομα ε, διαπίστωσα ότι είχαν πολύ μεγάλες προσδοκίες από εμά ως εθνικές υπηρεσίες. Μάλιστα, οι προσδοκίες αυτές ε, μπορούν να συνοψιστούν σε δύο βασικούς ερωτήματα. Καταρχώς, ε, αν η υπηρεσία πουλά προϊόντα ή εμπορικά σήματα ή αν δίνουμε το έναυσμα για τη διεθνοποίηση και τη συνεργασία. Δεύτερον, η Εθνική Υπηρεσία είναι τράπεζα, λοταρία, διοίκηση ή είναι ένας εταίρος ε, για τα ιδρύματα που θέλουν να υλοποιήσουν ε, διεθνή προγράμματα. Τα ερωτήματα αυτά, στη συγκεκριμένη μας περίπτωση, επειδή ε, είχαμε μόνο την ε, βασική δράση 1 και 2, αλλά έχουμε και άλλες δράσεις όπως στο Erasmus+, ε, e-training και σχολική εκπαίδευση, έχουμε και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και το ΙΠΑΛ e και προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούμε να τα συγκεράσουμε όλα αυτά. Δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω. Τα συμπεράσματά μας ήταν ότι καταρχάς πρέπει να λάβουμε υπόψη τι πρέπει να κάνουμε βάσει και του Erasmus Plus, αλλά δεν αφορεί μόνο τα χρήματα το θέμα αυτό, αφορά και τη διεθνή διάσταση. Και πρέπει να εξηγήσουμε ότι αυτά όλα πρέπει να είναι εφικτά. Μην αφήσετε να σας παραπλανήσουν τα χρήματα και οι δυνατότητες. Δεύτερον, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις ε, ομάδες στόχο που έχουμε και το, από πού ξεκινάνε τα, αυτά θα τα παραλείψω. Πάμε τώρα στη δομή. Ε, λάβαμε υπόψη μας δύο αρχές. Έγινε η μετάβαση από μια προσέγγιση ανατομέα και αναπροϊόντος σε διαχείριση λογαριασμών και στην διεθνοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση λογαριασμών δεν ε, προωθείται τον Γκρούντιχ, τον Λεωνάρντο κλπ. Υπάρχει μια ομάδα συμβούλων που όλοι έχουν ένα κλάδο πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέσσερις ανθρώπους έχουμε, μην φανταστείτε ότι έχουμε και 200 σε μια αίθουσα, μικρή υπηρεσία είμαστε υπάρχει κάποιο ο οποίο είναι ειδικό στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι στο ε, ομάδα στόχο 1 και 2. Πηγαίνει στα σχολεία και ρωτάει τι ιδέε έχετε, τι φιλοδοξίε έχετε και μετά προσπαθούμε να βρούμε τον καταλληλότερο τρόπο να ξεκινήσει αυτή η διεθνή διάσταση. Το ίδιο γίνεται με την ανώτερη εκπαίδευση και το ίδιο γίνεται και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε συνδυασμό με την αργοργασία και την ε, εκπαίδευση των ενηλίκων σε συνδυασμό με τι δημόσιε αρχέ και πρέπει να ξέρουν όλο το πρόγραμμα, να μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, γιατί στη δομή του προγράμματος, κυρίως στη δράση 2, ε, το γεγονό ότι είναι κάποιο σχολείο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει αίτηση για τη σχολική εκπαίδευση στη δράση 2. Γι' αυτό ακριβώ επιλέξαμε να έχουμε διαχείριση λογαριασμών και παροχή συμβουλών. Κάποιε συστάσει, πολύ σύντομα, θα σταθώ στι πιο σημαντικέ, όχι επειδή είμαι διευθυντή μια εθνική υπηρεσία, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε το ρόλο των ε, εθνικών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι υπάρχουν πολύ μεγάλε προσδοκίε όσον αφορά την παροχή συμβουλών. Να έχουμε ε, ιδέες ε, σε καλά προγράμματα, διότι υπάρχουν πολλέ ιδέε ε, και βγαίνουμε από μια μακρά περίοδο που προσπαθούσαμε να έχουμε διαβίω βάθηση και εράσμου πλά μαζί και τώρα πλέον έχουμε το περιθώριο να αρχίσουμε να εργαζόμαστε με τον κλάδο, εντό του κλάδου και όχι απλώ να εφαρμόζουμε διοικητικές ε, ε, διαδικασίε, να είμαστε εταίροι στα προγράμματα πράγματα. Κάποιες προτάσεις για τον προπολογισμό. Τα διάβασα και στις εκθέσεις αυτά. Υπάρχει μια γραμμική εξέλιξη. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μια όθηση και να δίνουν τα χρώματα λίγο πιο γρήγορα. Τώρα, για τις εθνικές υπηρεσίες έχουμε την ίδια γραμμική αύξηση της ε, ε, διαχείρισης και το κόστος της, αλλά τώρα όλα αυτά πρέπει να είναι έτοιμα σε τέσσερα χρόνια. Ως Εθνική Υπηρεσία λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σε θέση να επενδύσουμε τώρα σε κάποιους πόρους και κάποιες αρμοδιότητες και όχι μέχρι το 2020 όταν θα έχει αυξηθεί ο προπολογισμό. Και μια τελευταία σύσταση. Είναι πολύ δύσκολο από χρονική σκοπιά. Λάβαμε ένα πρόγραμμα εργασία το οποίο το ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον προπολογισμό το Σεπτέμβριο τα προγράμματα πρέπει να υποβληθούν το Φεβρουάριο την επόμενη χρονιά, που σημαίνει ότι έχουμε τέσσερι μήνε για να αντιμετωπίσουμε πιθανέ αλλαγέ. Και οι αλλαγέ αυτέ και η μετάφρασή του ε, στα του κλάδου είναι πολύ σημαντικέ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασία και προπολογισμό νωρίτερα, ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στι δομέ μα και στην επικοινωνία μα. Για την πληροφορική ούτε να την ακούω εναρμόνιση υπήρχαν κάποιες δυνατότητες και νομίζω ότι αυτό δεν έχει σχέση με τον επανασχεδιασμό του προϊόντος, αφορά τις ε, προκλήσεις ε, των Εθνικών Υπηρεσιών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάσουν τις πολύ μικρές προσαρμογές που πρέπει να γίνουν που θα έχουν σημαντικά αποτελέσματα. Και το συμπέρασμα το 2016 αλλά και στη συνέχεια σταθεροποίηση σας παρακαλώ, δώστε μας τη δυνατότητα να γίνουμε περισσότερο επαγγελματίε, δώστε μια αύξηση στο Erasmus Plus και τώρα έχουμε μια αύξηση στον προπολογισμό και πλέον θα έχουμε τις πρώτες τελικές εκθέσεις να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θα ε, γιορτάσουμε 30 χρόνια του Οράσμου του χρόνου και αν υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση για εκβάθρον αλλαγή του προγράμματο, έχετε κατά νου το 2020. Μην τα αρχίσετε τώρα γιατί θα πρέπει να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Ευχαριστώ. Many, many thanks. Uh, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ και για τις προτάσεις σας και για τα συμπεράσματα. συνδυάσατε τις συγκεκριμένες εμπειρίες από την καθημερινή ενασχόλησή σας με τα θέματα αυτά και ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Θα δώσω τώρα το λόγο. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος Βερ θέλει να μιλήσει τώρα ή αργότερα. Λιμπάτσκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε μια ερώτηση. Μια ερώτηση η οποία ε, προέκυψε σε ό,τι αφορά την παρουσίαση του τελευταίου ομιλητή. Τα εθνικά ιδρύματα, οι εθνικές υπηρεσίες ε, θα πρέπει να έχουν ένα εθνικό χαρακτήρα, θα πρέπει να προωθούν τη διεθνοποίηση. Σε ό,τι αφορά το Erasmus Plus τώρα, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει και μία ορισμένη εικόνα, αν θέλετε. Τρία χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό το γνωστό πρόγραμμα. Κατά δεύτερον, το Erasmus Plus είναι ε, ιδιαίτερο, ακριβώς επειδή είναι τόσο επιτυχημένο. Δεν έχουμε τόσες πολλές πρωτοβουλίες ε, ορόσημα, θέλετε, που έχουν στεφτεί με τέτοια επιτυχία. Και τρίτον, μια και περνάει η κρίση η ευρωπαϊκή μα ταυτότητα, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα προβλήματα αυτά με νέο μάτι, γιατί ενδεχομένω να μας βοηθήσουν τα ζητήματα αυτά για να δημιουργήσουμε μια γενιά πραγματικών Ευρωπαίων με ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και αυτό θα ε, μπορούσε να έχει σχέση και με την παρουσίασή σας και οι δύο στόχοι λοιπόν θα μπορούσαν να συμφιλειωθούν κατά από, την, ε, από το σήμα κρατεθένα, θέλετε του Erasmus Plus και θα πρέπει να απευθύνει την πρωτοβουλία αυτή σε όσο πιο πολλούς γίνεται και τώρα θα ήθελα να επικεντρωθώ στις πιο σημαντικές ιδέες τις οποίες ακούσαμε από κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου που διοργάνωσε η ομάδα μου, η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ένα επιχείρημα το οποίο το ακούσαμε επανειλημμένα Ενδεχομένω να μην συνάπτει τόσο πολύ με την εικόνα που έδωσαν οι εθνικές υπηρεσίες. Και για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Βάσει των δεδομένων, το Erasmus Plus δεν φαίνεται να είναι ένα καθολικό πρόγραμμα, δεν απευθύνεται σε όλους. Οι βασικοί δικαιούχοι είναι αυτοί που έχουν ουσιαστικά την οικονομική υποστήριξη των γονέων τους. Γιατί υπάρχουν ε, υποτροφίες, αλλά σε γενικές γραμμές ε, δεν αρκούν για να τα βγάλει πέρα κανείς χωρίς την βοήθεια των γονιών του. Οι υποτροφίες μπορεί να είναι διαφορετικού ύψους και αυτές οι διαφορές επίσης είναι πολύ μεγάλες. Και αυτό είναι προβληματικό. Και επίσης ε, η προσέγγιση στο θέμα των υποτροφιών διαφέρει. Για παράδειγμα, η Γερμανία έχει μειώσει 80% τις αποζημιώσει αυτές για όλους τους ε, ασκούμενους. Η Νορβηγία ποτέ δεν θα έκανε κάτι παρόμοιο. Και αυτά είναι τα δύο άκρα που σας ανέφερα. Σε ό,τι αφορά την ε, αναγνώριση του συστήματος CTS τώρα. Να πούμε ότι σπάνια να γνωρίζετε αυτό που πετυχαίνει κανείς σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, στο δικό του πανεπιστήμιο της χώρας του. Είναι απογοητευτικό αυτό και είναι πραγματικά λυπηρό που δεν μεταφέρονται αυτές οι μονάδες. Επίσης επιβάλλονται και κάποιοι φόροι σε κάποιες περιστάσεις, σε περιπτώσεις ε, και κάποια τέλη σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή τέτοιων νέων φοιτητών και νέων ακαδημαϊκών, νέων ερευνητών. Υπάρχουν λοιπόν πολλά εμπόδια τα οποία παρακολύουν την όλη διαδικασία. Η διαδομεακή κινητικότητα επίσης θα έπρεπε να προωθηθεί. Οι φοιτητέ ε, δεν είναι απαραίτητο, ξέρετε, να πάνε σε πανεπιστήμια. Μπορούν να κάνουν τη μαθητεία τους και την κατάρτισή τους σε επιχειρήσεις, σε εταιρείε. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο διαρκώς ε, παρουσιάζεται αφορά τις βασικές δυσκολίες σε ό,τι αφορά την διαθεσιμότητα κατανοητών πληροφοριών σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ξέρετε, ερμηνεύεται διαφορετικά. Με διαφορετικό τρόπο από ότι τα πανεπιστημιακά προσόντα. Ε, και θα ήθελα, επειδή πρέπει να κλείσω, και την εισηγήσή μου να κάνω δύο καταληκτικά σχόλια. Η δεύτερη βασική δράση. Εδώ θα πρέπει να δείξουμε προσοχή. Οι δράσει αυτέ που έχουν να κάνουν με την κοινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών θα έπρεπε να μας επιτρέψουν να αναδείξουμε και τη νέα γενιά δικαιούχων του Ορίζοντα 2020. Αλλά δεν είναι αρκετά υψηλό ο αριθμό, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ περίπλοκε οι διαδικασίε. Αυτό τουλάχιστον μου λένε. Οι εθνικέ υπηρεσίε θα πρέπει να συνεργαστούν. Αυτό ναι, υπογραμμίστηκε. Αλλά και κάτι άλλο που θα πρέπει να τονίσουμε. Η αποκέντρωση. Καθιστά τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα για τι εθνικέ υπηρεσίε. Για τι υπηρεσίε που σε γενικέ γραμμέ έχουν την έδρα του στι Βρυξέλλε. Η υπηρεσία των Βρυξέλλων ζήτησε αύξηση του προπολογισμού τη, αλλά η αύξηση των πόρων ήταν μάλλον επαρκή. Μία ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον ε, προπολογισμό. Τι θα γίνει με την στρατηγική για την κοινωνική συμπερίληψη και την ε, πολυμορφία τη νεολαία σύμφωνα με το Erasmus Plus. Τι θα γίνει με την στρατηγική αυτή θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη και άλλε εκπαιδευτικέ ανάγκε σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Προσβλέπω στη συνεργασία με τον κύριο Σβέρ, γιατί έχουμε συνεργαστεί μαζί και για την δίκαια στην Πολωνία. Ευχαριστώ. Ήμουν γενναιόδερη, γιατί διατελέστε και υπουργό παιδεία στη χώρα σα και για το πάθο σα, ο κύριο Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ που παρουσιάσατε τη μελέτη αυτή. Νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη για μας. Πρόκειται για μια μελέτη άρτια, αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό. Ως ευρωβουλευτές ε, μας προσεγγίζουν διάφορες οργανώσεις και πολίτες θέλουν να μοιραστούν μαζί μας το πρόβλημά τους, επομένως βλέπουμε σαφέστατα ποια είναι τα προβλήματα. Υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε σχέση με το Erasmus Plus. Λένε ότι είναι περίπλοκο, ιδίως όταν κάποιος θέλει να κάνει αίτηση για το πρόγραμμα και οι πολίτες θεωρούν ότι δεν υπάρχει ε, δυνατότητα επαρκούς πρόσβασης. Το Erasmus Plus είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα το οποίο έχει μεγάλη επιτυχία, το γνωρίζει ο κόσμος, είναι πολύ ε, ε, ελκυστικό, προσφέρει μεγάλες ε, δυνατότητες και αναπτύσσει και δεξιότητες για τους νέους ανθρώπους, κυρίως αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν με την εκπόδευσή τους. Και φυσικά το σχολείο και η διαβίου μάθηση είναι ένα απόσπαστο τμήμα της επιτυχίας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχουν εκθέσεις εφαρμογή και θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις διαδικασίες, όλες τις πρακτικές για να δούμε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Η αλλαγή χρειάζεται χρόνο και αν θέλουμε να αλλάξει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι αποτελέσματα θα προσκύψουν. Οι εθνικέ υπηρεσίε διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο και σίγουρα πρέπει να γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Αυτό θα προωθήσουμε άλλωστε και θα προσπαθήσουμε να άρουμε τα προβλήματα το συντομότερο δυνατόν. Ε, νωρίτερα σήμερα αναφέρθηκα στον προπολογισμό και είπα ότι χρειαζόμαστε αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και όχι απλώ αύξηση του προπολογισμού και αυτή τη δήλωση θα ήθελα να την επαναλάβω και εδώ. Χρειαζόμαστε ένα πάρα πολύ καλό μηχανισμό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Σβεντρόβα. Μετά θα σας κάνω μια ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ. θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στην ερώτηση ποιος είναι ο ρόλος των εθνικών γραφείων, των εθνικών υπηρεσιών για το Εράσμος. Απλά να ενημερώνουν, ε, να διαχειρίζονται, να αποστέλνουν ε, αξιολογήσεις για, τα, για ό,τι έχει προηγηθεί. Είναι πολύτιμη φυσικά η ε, συνεργασία τους. Βέβαια τα στοιχεία για τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση δεν είναι επαρκή. Υπήρχε ένα πρόγραμμα στα πλαίσια των κομβικών δραστηριοτήτων υπαριθμών 2 από κάποια πανεπιστήμια. Τέσσερις μήνες μετά το πανεπιστήμιο δεν γνωρίζει ακόμα αν έχει γίνει δεκτή η πρόταση και αν θα χρηματοδοτηθεί στην περίοδο 16-17 τέτοιου είδους ε, θα έλεγα ε, καθυστερήσεις ε, είναι αρνητικές. Αν τα πανεπιστήμια αυτά με τέτοιου είδους χρόνους που απαιτούνται δεν προλαβαίνουν να προετοιμαστούν σωστά. Έχουμε λοιπόν και τέτοιου είδους αρνητικές θα έλεγα εμπειρίες. Νομίζω ότι το σύστημα εδώ δεν λειτουργεί σωστά. Είναι σαφές ότι απαιτείται να υπάρξει απλοποίηση των κανόνων και όταν μιλάω για απλοποίηση των κανόνων δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στη συμπλήρωση των αιτήσεων αλλά και στον χρόνο τον οποίο θα πρέπει να περιμένει κανείς για να του δοθεί μια απάντηση για την αξιολόγηση από την οποία πέρασε. Ο χρόνος αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αρνητικά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα έχει το πρόγραμμα αυτό όταν και αν λειτουργήσει. Υπάρχει ένα πρόβλημα χρονισμού λοιπόν και καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σωστά τα ωφέλη από το παρόν σύστημα. Οι μελέτες που έχουν γίνει γύρω από αυτό είναι ενδιαφέρουσες, αλλά θα έλεγα τα τελικά συμπεράσματα είναι κάπως περιορισμένα και δεν υπάρχει απόλυτη, ε, απόλυτα πλήρης ενημέρωση. Ευχαριστώ για τις μελέτες αυτές, αλλά δεν γνωρίζω παρόλα αυτά αν η τσεχική ας πούμε εθνική υπηρεσία έχει πάρει σε αυτή την συνεννόηση και τη συνεργασία. Και αν το 2020 ας πούμε θέλουμε να αξιολογήσουμε το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, απαιτείται μια θα έλεγα ε, λεπτομερέστερη ανάλυση των ισχυρών και των ε, μη ισχυρών σημείων των μηχανισμών σε εθνικό επίπεδο απαιτείται να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις αλλαγές οι οποίες θα είναι χρήσιμες και να προετοιμαστούμε έτσι σωστά και για τη νέα περίοδο μετά από το 2020. Ήδη έχουμε ξεκινήσει λοιπόν να εμβαθύνουμε στο θέμα και δίνω τον λόγο στον κύριο Μόρκανο. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, αλλά έχω την, σχέση, θέση ότι σε σχέση με τα νέα προβλήματα της Ευρώπης, την προστασία της δημοκρατίας, την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών είναι κάτι το οποίο σε επίπεδο πολιτισμικό θα πρέπει να φροντίσουμε, να κυδαιμονεύσουμε αν θέλετε, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην καταπολέμηση της ριζοπαθικοποίησης. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι θέματα ε, τα οποία θα πρέπει να δούμε και μέσα από το σημερινό μας αντικείμενο συζήτησης. Πρέπει τέτοιου είδους προγράμματα να υποστηριχθούν ιδιαίτερα στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών και αναφέρομαι εδώ στις ΜΚΙΟ που ασχολούνται με τη νεότητα. Και μια, αν θέλετε, συμπληρωματική ερώτηση. Η αύξηση η οποία προβλέπεται για το Erasmus Plus για τους νέους είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι ότι είναι θετικό. Μέχρι τώρα όμως έχει εν μέρη αποδειχθεί αποτελεσματικό. Γιατί? Γιατί το σημαντικότερο τμήμα της αύξησης αυτής προβλέπεται για το 2017 και μετά. Ως εκ τούτου λοιπόν αντικειμενικά έχει υπάρξει μια κάποια στασιμότητα στις λειτουργικές πιστώσεις. Σχετικά τώρα με την έλλειψη των πόρων και σε ποιο βαθμό η έλλειψη αυτό, αυτή των πόρων έχει εμποδίσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να παίξουν τον ρόλο τον οποίο καλούνται να παίξουν. Θα πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε εμείς στον τρόπο συνεργασίας μας με την κοινωνία των πολιτών. Αν δεν λάβουμε υπόψη την κοινωνία των πολιτών στις σχέσεις της με τα θεσμικά όργανα θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Τρούπελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλες τις παρουσιάσεις. Να τονίσω ότι συμφωνώ με κάποιες από τις συστάσεις και κάποια από τα πορίσματα. Ασφαλώς δεν είναι εντελώς καινούργια, αλλά έχουν την ίδια εφαρμογή σε ό,τι αφορά την ευελιξία, τη μεγαλύτερη ευελιξία στα πλαίσια του προπολογισμού, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς πόρων από το ένα τίτλο από το ένα κομμάτι των άλλων. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ε, δικαιούχους και τους υποψηφίους. Μας μίλησαν λοιπόν ε, υποψήφοι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια νέα πλατφόρμα και θα μπορούσαμε πολλά να κάνουμε για να βελτιώσουμε το πρόγραμμα και να υπάρχει καλύτερη διαχείριση και του προγράμματος. Και μια ερώτηση έχω να σας κάνω. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τους τίτλου των παλαιών προγραμμάτων, είπατε ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε και στα άτομα που παραδοσιακά ενδιαφέροντουσαν για τα προγράμματα αυτά. Εσείς είπατε, κύριε Τρατσφέρτ, ότι πρέπει να στραφούμε σε νέους, ε, σε νέε ομάδε στόχου. Τι θα γίνει λοιπόν, πώς θα ενημερώνουμε για τα νέα ονόματα των ε, προγραμμάτων, γιατί ως τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς μας λένε ότι θα πρέπει να αναγνωρίζετε το πρόγραμμα από το όνομα το παλιό, προκειμένου να υπάρχει μια συνέχεια. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να μας προτείνετε κάτι γιατί να κάνουμε στο μέλλον σε ό,τι αφορά τις ονομασίες των προγραμμάτων. Ωραία, τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο της αρμόδιας υπηρεσίας, τον Τμήματιάρχη τον Φιλίπ Βαντέλε. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιον από την εκτελεστική υπηρεσία, παρόλο που υπήρξαν ερωτήσεις ε, που απευθύνονταν προς αυτούς. Ελπίζω να λάβουμε απαντήσεις κάποια στιγμή. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Μισό λεπτό. Πιθανές ε, συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις, απαντήσεις μάλλον σε ερωτήσεις. Ε, θα δούμε αν μπορούν να απαντήσουν οι ομιλητές μας και μετά θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Σβέρ. Επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω για την παρουσία της εδώ μια ομάδα φιλοξενουμένους της κυρίας Γκυγιόμ. Έχουμε 7 εμπειρογνώμονες από την Πουργκίνιο που ασχολούνται με τον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της διαβίου μάθησης. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Χαιρόμαστε που σα έχουμε. Η Κομισιόν παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για την πολύ, ευχαρι... για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και για τις παρουσιάσεις των εθνικών ε, υπηρεσιών πραγματικά είναι πάρα πολύ ωφέλιμες και προφανώς μας βοηθάτε ιδιαιτέρως για να βελτιώσουμε το τρέχον πρόγραμμα Erasmus Plus γιατί αν ναι, ένα πράγμα είναι σαφές είναι ότι χρειάζεται βελτίωση. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αποτελεί ενδεχομένω το πλέον επιτυχημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ότι η αξιολόγηση στο τρέχον κλίμα, στην τρέχουσα ατμόσφαιρα, χρειάζεται πιο πολύ παραποτέ. ποτέ. Κοιτώντας λοιπόν και τι έχει γίνει στο παρελθόν, πιστεύω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει μεγάλο, μεγάλη πρόοδο και την επόμενη χρονιά θα α, γιορτάσουμε την 30η επέτειο του ράσμους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσει, και αντίτρα με το Συμβούλιο που δεν έβλεπαν γιατί θα έπρεπε να υπάρχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση ε, με πολύ περιορισμένη χρηματοδότηση αρχικά και τώρα 30 χρόνια αργότερα έχουμε ένα πολύ εύρωστο πρόγραμμα με εύρωστη χρηματοδότηση που συνενώνει τις στόχους της εκπαίδευσης και της νεολαίας και αποτελεί το πιο γνωστό πρόγραμμα σε 28 χώρες και στις 28 χώρες. Και επίσης νομίζω ότι αναφέρθηκε και στην ε, έκθεση πρόκειται για ένα βήμα πολύ σημαντικό για την πρόοδο του Erasmus Plus. Έτσι πιστεύουμε και εμείς. Τώρα πια ε, επτά ε, επιμέρους προγράμματα ενώνονται κάτω από την ομπρέλα ενός προγράμματος. Και θεωρούμε ότι το Erasmus Plus ε, έχει πετύχει αποτελέσματα. Και τι έχουμε πετύχει ως τώρα. Χάρη στο πρόγραμμα, πάνω από 2 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν ωφεληθεί από μία περίοδο κινητικότητα στο εξωτερικό. Μιλάμε για 2,3 εκατομμύρια συμμετέχοντες που έχουν ενεργά συμμετέχει στο πρόγραμμα. Χάρη στις εθνικές υπηρεσίες και το εκτελεστικό γραφείο έχουμε χρηματοδοτήσει 50.000 προγράμματα, έργα μάλλον, ε, συνενώνοντας ε, και κάνοντας να συνεργαστούν 175.000 ε, υπηρεσίες. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε περαιτέρω το Erasmus Plus γιατί ξέρουμε ότι αυτό απασχολεί το Κοινοβούλιο και βλέπουμε ότι 37% είναι άτομα από μειονεκτικές, από μειονεκτικό κοινωνικό υπόβαθρο. Επίσης έχουμε ασχοληθεί με το θέμα των ε, αποζημιώσεων, των ε, υποτροφιών, οι οποίες ομολογμένως είναι χαμηλές και προσπαθούμε σε άτομα χαμηλής ε, μισθολογικής προέλευσης να δώσουμε ένα τόπο από 100 ευρώ και για τους φοιτητές. Και επίσης για πρώτη φορά κάνουμε τη διάκριση μεταξύ κόστου διαβίωσης στην χώρα προέλευσης και στη χώρα υποδοχής προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν επαρκή χρήματα για να μπορέσουν να ζήσουν στη χώρα υποδοχής. Επίσης, βλέποντας τι γίνεται, τι γίνεται με τους φοιτητές υψηλής εξειδίκευσης και υψηλής εκπαίδευσης, βλέπουμε ότι είναι πιο μεγάλο το ποσοστό των μειονεκτικών ε, ε, φοιτητών μεταξύ αυτών. Και πραγματικά βλέπουμε 100% πλήρη υλοποίηση κάθε έτος. Αυτό δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο πρόγραμμα. Είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση. Αυτό είναι ασφαλώ θετικό στοιχείο, αλλά προφανώς ε, σημαίνει και κάτι αρνητικό. Σημαίνει ότι κάθε χρόνο πολλά project υψηλής ποιότητας απορρίπτονται. 80% δηλαδή των ε, ετούντων απογοητεύονται για την αρνητική απάντηση και επίσης ο χρόνος αξιολόγησης σημαίνει, τι σημαίνει αυτό, ότι οι εθνικές υπηρεσίες πρέπει να δαπανούν πολύ χρόνο και κόπο για την αξιολόγηση πολλών ε, project, ενώ ξέρουν ότι θα μπορέσουν τελικά να χρηματοδοτήσουν ένα περιορισμένο μόνο ποσοστό αυτών. Κάτι άλλο το οποίο αποτελεί μεγάλη επιτυχία είναι η ευηλεξία του προγράμματος. Αυτό το παραδέχτηκε και το Συμβουλίο και ε, το Κοινοβούλιο. Να υπάρχει ένα πρόγραμμα με έναν στόχο. Και βλέπουμε ότι ξεκίνησαν διαπραγματεύσει το 2011 και τα ολοκληρώθηκαν το 2013 και έκτοτε έχει αλλάξει το συγκείμενο το πολιτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε το μεταναστευτικό, η ανάγκη επενδύσεων για την κοινωνική, την κοινωνική συμπερίληψη, την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, την ατζέντα για τις νέες, ε, τα νέα προσόντα της Επιτροπής και για όλα αυτά τα θέματα καταφέραμε να μετατοπίσουμε τις προτεραιότητες του προγράμματος και για τα, τις νέες ε, ανερχόμενες ανάγκες. Κάτι που αναφέρθηκε επίσης και είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όταν μιλάμε για τις δυσκολίες της υλοποίησης, της, την εκτελεστική υπηρεσία και τις εθνικές υπηρεσίες που το 2014 και 2015 είχαν πραγματικά ε, έκαναν τιτάνιο έργο για να ολοκληρώσουν όλα τα, όλες τις διαδικασίες, όλα τα συστήματα τα απολογιστικά και τα IT και παράλληλα ξεκίνησαν και άνοιξαν καινούργια συστήματα και καινούργιες διαδικασίες, οι οποίες δεν ήταν πάντα ομολογουμένω πολύ επιτυχημένε. Αλλά θεωρούμε λοιπόν ότι συνολικά βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, το οποίο και κάτι άλλο το οποίο ακούσαμε στη διάρκεια της συζήτηση το επίπεδο αναγνώρισης. 85% των ε, μονάδων που ε, πετυχαίνει κανείς ε, στο εξωτερικό αναγνωρίζονται στην μεταπή στην πατρίδα του. Και περιμένουμε το ποσοστό αυτό να αυξηθεί σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των δεκτικών μονάδων. Γιατί θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης αυτής. Είμαστε σχεδόν, ε, αν θέλετε, στον δρόμο της πλήρους αναγνώρισης και είμαστε αισιόδοξοι γενικά. Ότι θα πετύχουμε και θα υπερβούμε και τους στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή του προγράμματος. Προφανώς ε, θα πρέπει, ωστόσο, να αντιμετωπίσουμε κατάματα τις πραγματικές προκλήσεις. Και ετέθησαν διάφορα ζητήματα και στη συνάντηση με τις εθνικές υπηρεσίες και με τους δικαιούχους. Και αν θέλετε να σας αναφέρω και τέσσερα ζητήματα, τα οποία αναφερθήκαν και στη συζήτηση σήμερα. Το θέμα του IT καταρχάς, αυτό αποτέλεσε πραγματική πρόκληση. Το να περάσουμε από 7 διαφορετικά προγράμματα με διαφορετικές διαδικασίες, με διαφορετικά εργαλεία, διαφορετικούς τίτλους, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, με ένα, μία ενιαία προσέγγιση και να αναπτυχθούν νέα εργαλεία IT από το μηδέν σε πολλές περιπτώσεις και σε κάποιες ε, περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που ονομάζονται εταιρικά εργαλεία. Κάποιοι δεν ταιριάζουν απαραίτητα στι ανάγκε ενό τέτοιου προγράμματο όπω το Erasmus Plus. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση λοιπόν και αναγνωρίζουμε τον εφιάλτη που πέρασαν οι εθνικέ υπηρεσίε το 2014. Ελπίζω όμως όλοι να συμφωνείτε ότι βαθμιαία και σταδιακά υπάρχει πρόοδος. Όλα αυτά συζητήθηκαν επισταμένως με τις εθνικές υπηρεσίες και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε και τα υπόλοιπα προβλήματα προκειμένου το αργότερο το, στα αρχές του 2017 να έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον IT. Και να προσθέσω στο σημείο αυτό ότι προφανώς οι δικαιούχοι θα τους πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να δουν τις αλλαγές αυτές. Προτού εφαρμοστούν και γίνουν αισθητέ πραγματικά οι αλλαγές και η πρόοδος, αυτό μπορεί να πάρει μήνες, μήπως και ίσως και χρόνια. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ένα άλλο θέμα το οποίο απαντάτε ε, τακτικά είναι οι μικρές οργανώσεις και πώς τις αντιμετωπίζουμε. Θεωρώ ότι στην αρχή δεν υπήρχε ισορροπία. Ήμασταν πιο πολύ εστιασμένοι στα μεγάλα project. Εν τω μεταξύ έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα και επιλέγονται και μικρή κλίμακα project. Στι ε, αιτήσει λοιπόν το 2016 βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ πιο πολλέ ε, αιτήσει από μικρέ οργανώσει για μικρά project. Αυτό είναι ενδιαφέρον και νομίζω ότι επιτυχάνει μεγαλύτερη ισορροπία. Ένα άλλο θέμα. Το θέμα των brand names, των ε, επωνυμιών που έχει χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενη γενιά. Εδώ διαπιστώνουμε ότι η πρόθεση του Erasmus Plus έχει ωφέλη για την διατομεακή επίδραση του προγράμματος, γιατί θέλουμε να υπάρχουν πιο πολλές οργανώσεις νεολαίας για να συνεργάζονται με τα σχολεία, με τα ιδρύματα της και άνω της Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η μεγαλύτερη διασύνδεση. Και θα πρέπει επίσης να προσελκύσουμε και νέους δικαιούχους. Και το γεγονός ότι γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του Εράσμους και η προσέγγιση ότι θα εξηγήσουμε το Erasmus στο Erasmus Plus θα είναι μια ευκαιρία να εξηγήσουμε και τα θέματα επωνυμίας. Και τέλος, να πω και δύο λόγια για την απλοποίηση. Να σας πω ότι τίποτα δεν είναι πιο περίπλοκο από την απλοποίηση. Αλλά να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε και περαιτέρω μέτρα. Για την χρηματοοικονομική λοιπόν υποστήριξη κάνουμε και άλλα βήματα για τις συμβάσεις. Έχουμε αναθεωρήσει τις συμβάσεις μεταξύ των εθνικών αρχών και των δικαιούχων και εκεί ελπίζουμε ότι θα μειωθεί το γραφειοκρατικό άχθο και τέλο για τι αιτήσει. Πάρα πολύ δύσκολο θέμα γιατί χρειάζεται μια σωστή εκτίμηση και αξιολόγηση των ε, αιτήσεων. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε κάποιε πληροφορίε για τι αιτήσει. Αλλά παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να μειώσουμε τον αριθμό των ερωτήσεων και την έκταση των αιτήσεων. Και ακόμα αυτό θα συμβεί ήδη από το 2017. Μην σα πω ότι καταρτίζουμε και online τέτοιε αιτήσει για να διευκολύνουμε περαιτέρω την κατάσταση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και εδώ κλείνω. Sorry. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, αλλά ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος, γιατί πρέπει να απαντήσει και ο συνάδελφος Βέρ. Να πω κι εγώ δύο λόγια όμω πρώτα. Θέλετε να απαντήσετε όλοι ή κάποιοι από εσά. Όπως και να έχει ένα λεπτό θα έχετε. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε χρόνο. Πέντε ώρα πρέπει να τελειώσουμε. Yes, the name. Ναι, τα ονόματα. Αυτό είναι ένα σύστημα, ε, ε, θέμα το οποίο ανακύπτει συνεχώς. Δυστυχώς δεν μπορεί να βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Καταλαβαίνω όλους αυτούς που λυπούνται διότι υπήρχε μια ταυτότητα, δεν ξέρω, σαν την Κρούντιχ. Και τώρα θέλουν, ε, πρέπει να τη χάσουν, υπάρχει και για τις ονομασίες, ε, ε, μπορεί να πρέπει κάποιος να λάβει ένα τελείως καινούριο όνομα. Για τη διαβίου μάθηση, για παράδειγμα, εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε, είναι πολύ τεχνικός όρος. Το Εράσμους 1, ε, εντάξει, κέρδισε το Εράσμους, δεν μπορούν να κερδίσουν όλοι. Ε, θεωρώ ότι σε ένα πρόγραμμα που λέμε ότι κυρίως μας ενδιαφέρουν οι δραστηριότητες, δεν ασχολούμαστε τόσο με τους τομείς, είναι πολύ λογικό να υπάρχει μια κοινή ονομασία και να μην είναι τόσο ισχυρές οι επιμέρους ταυτότητες. Μια υπηρεσία είπε ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εννοεί στα σοβαρά, τότε πρέπει να αναδιοργανωθεί δεν μπορείτε να έχετε ένα τμήμα για την ανώτατη εκπαίδευση, θα πρέπει να έχετε ένα τμήμα για την κινητικότητα. Τέλος πάντων, μακρηγόρησα. Παρακαλώ, υπόλοιποι. Θα ήθελα να πω ότι η μεγαλύτερη χρηματοδότηση δεν είναι απαραίτητη μόνο για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα ή την αποδοτικότητα των προγραμμάτων ε, του Erasmus Plus και των έργων, αλλά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τις δραστηριότητες και τη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών. Πρέπει να ορίσουμε ποιες είναι οι καινοτομίε. Πρέπει να υπάρξει μια νέα και βελτιωμένη διαδικασία, νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχουμε στις οργανώσεις των πελετών μας και χρειαζόμαστε λιγότερο γραφειοκρατικό άχθος. Πρέπει να υπάρχουν εργαλεία ενημέρωσης και πάρα πολλές βελτιώσεις στην εφαρμογή του προγράμματος Εράσμους για να βελτιώσουμε και την ε, αποτελεσματικότητα των ε, ε, προγραμμάτων. Ευχαριστώ, κύριο κύριος ένα μικρό σχόλιο. Οι μικρέ οργανώσει σίγουρα χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη. Είναι σαφέ ότι η τάση πηγαίνει από τι μικρότερε προ τι μεγαλύτερε οργανώσει που είναι πιο έμπειρε, που έχουν περισσότερου πόρου κ.ο.κ. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να υπάρχει περιθώριο ώστε οι μικρότερε οργανώσει να αντιμετωπίσουν και αυτέ το πρόγραμμα. Αυτό είναι βέβαιο εξαρτάται από την μορφή που προσφέρουμε αλλά και από την παροχή υπηρεσιών από τις ε, ε, εθνικές υπηρεσίες. Εμείς λοιπόν είμαστε διαμοσολαβητές, αυτοί που διευκολύνουμε όπως ακούστηκε ήδη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλοι ε, βρίσκουμε το δρόμο μας και όταν αναφερόμαστε σε ιδιαιτερότητες ενός τομέα δεν αφορά μόνο την ονομασία αυτό Χρειαζόμαστε να χρησιμοποιείτε το όνομα στην πράξη για να αναγνωρίζετε και ως όνομα. Χρειαζόμαστε όλη την υποστήριξη των εθνικών υπηρεσιών και υπάρχει διαφορετική προσέγγιση σε κάθε χώρα γιατί είναι τελείως διαφορετική και η νοοτροπία. Δεν μπορούμε να έχουμε μία προσέγγιση και είμαστε ενωμένοι εν την ποικιλομορφία μας και αυτό νομίζω ότι ισχύει και για το πρόγραμμα. Τελευταία παρατήρηση παρακαλώ. Αντιλαμβάνομαι και πολύ συχνά ακούω στον τομέα των νέων ότι ο τίτλος Youth in Action αξίζει τον κόπο και συμφωνώ, διότι το Youth in Action για μένα δεν είναι ονομασία, είναι η βάση του Erasmus Plus που λέει ότι το Erasmus Plus έχει κάτι να προσφέρει στους νέους. Δεν είναι η Άννα Φρανκ, επιτρέψτε μου λίγο την υπερβολή, όπως έχουμε την Γκρούντι, το Λεωνάρδο και το Erasmus και το Κομένιους. Αυτά δεν είναι βασικές γραμμές που λέμε ότι υπάρχουν ε, ε, προγράμματα για τα σχολεία. Είναι μια αναφορά σε ένα προηγούμενο πρόγραμμα το οποίο ήταν τελείως διαφορετικός. Ε, το να χρησιμοποιήσουμε εκ νέου αυτά τα ονόματα θα δημιουργήσει ανατορυχή και θα χαθεί και η σημασία του τομέα. Αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται και το βλέπουμε στο Erasmus Plus ε, είναι η κινητικότητα των φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση και αυτό που δεν έχουμε στο εθνικό πλαίσιο είναι ένας υπουργό παιδείας που να λέει ότι η κινητικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση, ναι, αυτό το λένε όλοι, αλλά είναι πολύ σημαντική και η κινητικότητα των βετεράνων να υπάρχει ένας ε, ε, δάσκαλος ο οποίος θα πάει ε, να παρακολουθήσει πώς κάνει τη δουλειά του κάποιος άλλος. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να δούμε λοιπόν όλες τις δυνατότητες του προγράμματος και όχι μόνο την ανώτατη εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τσφέρ να πω τρία πράγματα. Πρώτον, νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση είναι πολύ σημαντική στιγμή γιατί πλησιάζουμε στα γενέθλια του ε, Εράσμους πριν 30 χρόνια. Θυμάμαι την Κοράντι, μια Ιταλίδα η οποία ξεκίνησε τις ανταλλαγές ε, με την Ισπανία και σύν της άλλης έχουμε να γιορτάσουμε και τα 20 χρόνια της εθελοντικής προσφοράς. Εμείς λοιπόν, όπως έχουμε ήδη πει ε, και με τον Επίτροπο, θέλουμε ακριβώς την εθελοντική προσφορά να την εντατικοποιήσουμε ακόμα περισσότερο και να την αναζωογονήσουμε στο μέλλον. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι οι αθλητικές δραστηριότητες βέβαια. Και θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με τις στρατηγικές δράσεις, και τις εγκάρσιες στον τομέα της συνεργασίας, η συμμαχία της γνώσης, οι εταιρικέ σχέσεις. Ένα άλλο θέμα και μέσα στο Εράσμους. Είναι σαφές ότι πρέπει να χρησιμεύσουν όλα αυτά για να βελτιώσουν αυτό το οποίο ονομάζουμε ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο. Υπάρχει επίσης ε, το θέμα του Master Guarantee. Εδώ είναι κάτι το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά και θα πρέπει να δούμε γιατί. Υπήρξε ίσως ένας αποπροσανατολισμός των στόχων Ξέρετε ότι η λέξη Εράσμους είναι κάτι το πάρα πολύ καλό, αλλά σύν της άλλης λειτουργήσε από προσανατολιστικά, γιατί πολλοί θεώρησαν ότι αφορά μόνο στους φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με την ονοματολογία, είναι σημαντικά τα ονόματα και θα επανέλθουμε σε αυτό που είπε η κυρία Τρούπελ ε, θα πρέπει να πω ότι το μεγάλο καπέλο είναι το Εράσμους και μετά θα πρέπει να υπάρξει αναφορά σε διαφορετικά επιμέρους θέματα τα οποία δεν ταυτίζονται με τις πανεπιστημιακές σπουδέ. Ο συνάδελφος Σβέρ, νομίζω ότι η συνάντηση μέχρι τώρα ήταν πραγματικά χρήσιμη. Σας ευχαριστώ πολύ θα ήθελα και εγώ να παρουσιάσω κάποια από τα δικά μου συμπεράσματα, τα οποία νομίζω συμπίπτουν με τα δικά σας. Θα συμφωνήσω με τους τέσσερις προλαλήσαντες ομιλητές για σήμερα το απόγευμα. Έλαβα υπόψη τα σχόλια των συναδέλφων, επίσης τα δεδομένα τα οποία παρουσίασε ο καθηγητής κ. Βέχτερ νομίζω ότι λειτουργούν με θετικό τρόπο. Όταν συζητάμε θέματα με κάθε μία από τις εθνικές υπηρεσίες η αίσθηση την οποία έχουμε ε, είναι διαφορετική ίσως από χώρα σε χώρα. Γι' αυτό ακριβώς η μελέτη αυτή ε, είναι κάτι που αξίζει νομίζω να μελετηθεί και τα συμπεράσματά της ε, πρέπει να τύχουν της απαιτούμενης προσοχής. Υπάρχει επίσης η διαπίστωση ότι η διατομιακή συνεργασία βελτιούται, οι χρηματοδοτήσεις επίσης βελτιούνται, αλλά δεν πάβουν οι καθυστερήσεις να είναι σημαντικές. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό όσο δύσκολο και αν είναι κάτι τέτοιο. Έχουμε στείλει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σήμερα σε όλους όσους εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης. Υπήρξαν αρκετές και σημαντικές διαφορετικές άλλαγες. Θα μπορούσαμε να δώσουμε αν θέλετε και βραβείο Νόμπελ στον Επίτροπο που αποφασίζει να μην αλλάξει τη δομή του σύνολου συστήματος αλλά να μην ξεκινήσει δηλαδή από το μηδέν. Ξέρουμε ότι ορισμένες υπηρεσίες είχαν προβλήματα όταν ε, λειτουργήσαν μεταβατικά σε ένα νέο και πέρασαν σε ένα νέο μηχανισμό. Απαιτείται λοιπόν να έχουμε λιγότερα μέσα ίσως στη διάθεσή μας, αλλά τα οποία αυτά μέσα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά. Ελπίζω ότι το σύστημα θα παραμείνει σταθερό για αρκετό καιρό και δεν θα υπάρξουν νέες αλλαγές οι οποίες θα τρομάξουν τους χρήστες. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές υπηρεσίες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης, ιδιαίτερα την συνεργασία με την εκτελεστική υπηρεσία που ασχολείται με τα οπτικοακουστικά και εκπαιδευτικά θέματα και που έχει την έδρα της εδώ στις Βρυξέλλες. Εναρμόνιση λοιπόν, ναι, τυποποίηση λοιπόν, ναι, είναι καλά πράγματα. Όμως θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει και ένα επίπεδο επιθυμητό αυτονομίας και ευελιξίας. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω από τις παρουσιάσεις σας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης την συνεργασία ανάμεσα στις ίδιες τις εθνικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε σχέση με τα προγράμματα της νεότητας. Νομίζω ότι οι υπηρεσίες λοιπόν μπορεί να λειτουργήσουν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή τους επόμενους μήνες θα αναλύσουμε προσεκτικά τις μελέτες σας. Φυσικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε μία εβδομάδα να τις αναλύσει κανείς προσεκτικά και να αναλύσει όλα τα θετικά και τα αρνητικά τα οποία διαπιστώσατε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Υπάρχει επίσης ένα άλλο σημαντικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι δεν είναι κάτι το θετικό οι ε, μεγάλοι σε εισαγωγικά παίκτες να έχουν το πλεονέκτημα. Αυτό αφορά το σύνολο των οργανώσεων και το σύνολο των προγραμμάτων. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε επίσης και τους ε, μικρότερους σε εισαγωγικά παίκτες. Ως εκ τούτου το Erasmus Plus θα καταστεί επιτυχέστερο της ε, σημερινής του μορφής. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι το Erasmus Plus δεν έχει μόνο ένα τεράστιο δυναμικό βελτίωσης, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάστασης των νέων γενικότερα, αλλά έχει και την δυνατότητα να βοηθήσει ε, της εμπλοκής όλων των νέων σε δημοκρατικές διαδικασίες. Σημερίζομαι λοιπόν την τελευταία άποψη την οποία εξέφρασε ο κύριος Φέρ. Νομίζω λοιπόν ότι Περάσαμε δύο ώρες εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι αυτές οι εκθέσεις εφαρμογής θα συνεχίσουν σήμερα και αύριο και είναι μια καλή ευκαιρία για μας και ελπίζω και για τους συνομιλητές μας που ασχολείται με το 70 σχεδόν της 100 των προγραμμάτων έχουν τεράστιες εμπειρίες αυτές οι εθνικές υπηρεσίες. Ελπίζω ότι ο κύριος Βέρ μαζί με τους Σκιώδης έχει πάρα πολύ υλικό για να συνεχίσει τις εργασίες του. Κλείνουμε λοιπόν την σημερινή συνάντηση με την παρούσα μορφή. Αμέσω μετά έχουμε μια κοινή συνάντηση με την Επιτροπή Ήτρε. Σε πέντε λεπτά. Μείνετε εδώ παρακαλώ, θα μιλήσουμε για τις δημιουργικές και πολιτιστικές ε, βιομηχανικές δραστηριότητες.